εργασίας ανηλίκων. Θα δώσω το λόγο πρώτα στους συντάκτες. Ο κύριος Ιτελβελτέ πρώτα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα που συζητάμε σήμερα. Πρόκειται για τις ευρωπαϊκές αξίες. Ε, υποβάλαμε την προφορική ερώτηση και συντάξαμε και ένα κοινό ψήφισμα για το λιθουανικό νόμο που ισχυρίζονται ότι προστατεύει τους ανηλίκους. Όμως το αντίθετο κάνει ουσιαστικά συνάδελφοι, γιατί αυτός ο νόμος ε, οδηγεί σε άγνοια ενίσχυση των ταμπού, των στερεοτύπων και στιγματίζει ε, τους ε, νέους ε, ομοφιλόφιλους και αμφιφιλόφιλους θα αποκλειστούν, θα τους ασκηθεί πίεση ε, δηλαδή θα ασκηθεί πίεση ε, και εκφοβισμός σε αυτούς τους νέους που υποτίθεται προστατεύει ο λιθουανικός νόμος. Ε, γι' αυτό το λόγο, συνάδελφοι, υποβάλαμε αυτή την προφορική ερώτηση και χαίρομαι γιατί το καλοκαίρι ήδη ο Επίτροπος Μπαρό μας έστειλε μία επιστολή όπου εκφράζει την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση αυτού του νόμου και μας ανακοίνωνε ότι θα παρακολουθεί εκ του σύνδεγγυ στο θέμα και για να μεριμνήσει ούτως ώστε οποιαδήποτε λιθουανική ηλεκτρονική νομοθεσία συνάδει πλήρω με το κοινοτικό κεκτημένο και με τι ευρωπαϊκέ αρχέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να παρεμβαίνει μόνο όταν παραβιάζονται οι κανόνε τη αγορά, αλλά κυρίω όταν παραβιάζονται ε, οι ευρωπαϊκές αξίες. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη διακριτική μεταχείριση. Η κοινότητα είναι μια κοινότητα αξιών που ενστερνίζονται σίγουρα όλοι οι Λιθουανοί συμπολίτες μας και λέω συμπολίτες γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είμαστε. Τώρα σε σχέση με το ψήφισμα συνάδελφοι ζητώ τη ρητή υποστήριξή σας ε, και κυρίως για την τροπολογία που αποσκοπεί στην ένταξη μιας εμνίας ε, στην ε, υφιστάμενη, υφιστάμενες μάλλον οδηγίες για την καταπολέμηση διακριτικής μεταχείρισης. Το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε. Ζητώ υποστήριξη επίσης ε, για την αίτηση που υποβάλλουμε μέσω του ψηφίσματος. Ζητάμε από τον Οργανισμό δηλαδή, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εκπονήσει νομική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο λιθουανικό νόμο. Και τέλος, συνάδελφοι, Νομίζω μπορούμε να είμαστε περήφανοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν αύριο εγκριθεί αυτό το ψήφισμα γιατί θα ακουστεί η φωνή των κοινών αξιών της ευρωπαϊκή Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπε και η προλαλή σας, εδώ σχετικά με αυτή την νομοθεσία πρόκειται ε, για ε, ένα νόμο όπου αμφισβητείται όχι μόνο το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και ε, η ελευθερία των ατόμων που μπορεί να είναι αμφι αμφιλόφιλοι οι ε, λεσβίες ε, οι ομοφιλόφιλοι και που μπορούν να βλαβούν από την ομοθεσία αυτή αντί από τις, ε, από τις πληροφορίες οπότε μπορεί να κινδυνεύσουν να πάθουν κατάθλιψη να μην μπορούν να χαρούν ε, την ε, νεότητά του ε, και να υπάρξουν ακραίες τάσεις. Άρα η νομοθεσία αυτή παραβιάζει τα δικαιώματα και γι' αυτό ο κύριος Μπαρό μας είχε δώσει ήδη μία απάντηση τον Ιούλιο και άλλωστε οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των ομοφιλοφίλων και ε, λεσβίων ε, ε, μας έγραψε ότι ελέγχει το θέμα και θα απαντήσει χωρίς όμως να μας λέγουν τι έχει γίνει έναντι του Λιθουανικού Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο δεν έχουμε πληροφορίες διότι η προηγούμενη Επίτροπος δεν είχε αποδεχθεί αυτό το νόμο αλλά το Κοινοβούλιο επιμένει και ελπίζουμε ότι μέσω αυτού του ψηφίσματος μπορούμε να προχωρήσουμε και ε, να απευθυνθούμε και στην ε, Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να αποφανθεί διότι θα πρέπει ε, να πούμε στην Ευρώπη ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί η ζωή των ομοφιλοφίλων παιδιών μόνο επειδή ένας νόμος το απαγορεύει. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ταβάρες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο νόμος αυτός ο στόχο έχει την προστασία των ανηλίκων κατά της ομοφιλοφιλίας. Ε, τι σημαίνει όμως αυτό ότι αν θέλω εγώ να πάω σινεμά και να δω το Brock Mountain στο Vilnius ε, θα μου λέει μια ταμπέλα ότι δεν μπορώ ή ότι θα πληρώσω πρόστιμο μέχρι 1500 ευρώ λόγω των τροποποιήσεων ε, που θα οδηγήσουν στο νέο ποινικό κώδικα που συζητείται τώρα στο Κοινοβούλιο. Κάτι μου έκανε εντύπωση αγαπητοί συνάδελφοι. Μια ημερομηνία. 14 Ιουλίου 2009. 14 Ιουλίου είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε εδώ, νέα αυτή η θητεία, 220 χρόνια από τις ε, ευρωπαϊκές αρχές, ε, ελευθερία έκφρασης και ελευθερία ε, συγκέντρωσης διότι και αυτό τώρα κινδυνεύει στην ε, Λιθουανία που απαγόρευσε ας πούμε την Gay Pride. Έχουμε καθήκον, ιερό θα έλεγα, να υπερασπίσουμε αυτές τις αξίες. Και από αυτού πρόκειται. Δεν ξέρουμε από πού ξεκινάνε αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρουμε πάντα πού οδηγούν και πώς ε, καταλήγουν. Και τι σημαίνει αυτή η ιστορία κατά της διάχυσης της ομοφιλοφιλίας. Πού, στα σινεμά, στα βιβλία. Το Βίλνιους μάλιστα είναι και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και δικαίω. Αλλά όποιος έχει τέτοιου είδους ε, προνόμια έχει και ευθύνε. Και το Βίλνιους έχει την ευθύνη να είναι όχημα και φορέας των αξιών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, κάνω έκκληση υπέρ του ψηφίσματός μας και η Επιτροπή μας ε, ε, ανέφερε τις απόψεις της. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Κάσμαν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως ομοφιλόφιλος μπορώ να πω ότι είμαι υπερήφανος για τα λόγια των ε, συναδέρφων. Η πρόταση αυτή αποτελεί παράβαση του άρθρου 6 και της οδηγίας πλαίσιο για τις μη διακριτικές μεταχειρήσεις την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών ε, και εναντίον των διακριτικών μεχειρήσεων ε, κατά των ομοφιλοφιλών ε, και λεσβιών. Ποιος προστατεύει ποιον λοιπόν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το 1998 εισήχθη ένα παρόμοιο νόμο στο Ηνωμένο και αναγνωρίστηκε και τότε και αναγνωρίζεται και τώρα ότι συνέβαλε στην ομοφοβία, στι διακριτικέ μεταχειρήσεις Φαινόμενα που καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων. Η πρόταση καταδικάστηκε και από μη κυβερνητικέ οργανώσει, την Διεθνή Οργάνωση Ομοφυλοφίλων, την ε, Διεθνή Αμνηστία και άλλου. Επηρεάζει τους ε, ίδιου τους ομοφυλόφιλου, τους δάσκαλους, τους νέους που ε, έτσι έχουν μειωμένη πρόσβαση σε βιβλία, σε έργα τέχνης που δημιουργεί ένας ομοφυλόφιλος ο Πλάτωνας, ο Σέξπιρ, ο Όσκαρ Βάιλντ, ο Βουλτ Βίτμαν, ο Τένισι Βίλιαμς, ο Τσαϊκόφσκι, ε, ο Έλτον Τζον, η Μαρτίνα Ναυρατήλοβα στο τένις, όλα αυτά είναι απαγορευμένοι καρποί. Λέμε λοιπόν, μιλήστε, σκεφτείτε και δράστε γιατί πρέπει οι νέοι να κατανοούν τον κόσμο σε όλη του την ποικιλομορφία και να σέβονται το διαφορετικό. Το αγάπα των πλησίων σου δεν έχει λιγότερη σημασία σε αυτή την περίπτωση. Κανονικοί άνθρωποι είναι οι ομοφιλόφιλοι που έχουν ε, ε, ε, υποστεί τόσες διακριτικές μεταχειρήσεις όπου θεωρούνται, που θεωρείται ότι αποτελούν απειλή κατά της κοινωνίας αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία μας. Η κοινωνία μας κρίνεται, όλες οι κοινωνίες κρίνονται, όχι πώς μετα... για το πώς μεταχειρίζονται τις πλειοψηφίε, πλειοψηφίες, αλλά για το πώς μεταχειρίζονται τις μειοψηφίες. Ας παραπέμψουμε αυτό το επικίνδυνο νομοθέτημα στις ρωμαϊκές καλένδες. Ευχαριστώ. Η Υπουργό Μάλστρομ. Ε, Ευχαριστώ, αξιότιμοι βουλευτές. Αρχικά θα ήθελα να τονίσω ότι η ελευθερία έκφραση, η κατάργηση της διακριτικής ε, μεταχείρισης ε, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της γενετήσια ταυτότητα είναι η λύθη της δημοκρατικής μας ε, κοινωνίας. Εμείς, η κοινωνία μας βασίζεται σε διάφορες αρχές, σε διάφορες αξίες και όλοι πρέπει να τις ενστερνίζονται. Δεν ναι, μπορούμε να ζητάμε από άλλες χώρες να μην παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ εμείς ε, οι ίδιοι δεν τα σεβόμαστε. Οι βασικές ελευθερίες, συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης, ε, προβλέπεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης και έχουμε και τα άρθρα 10 και 14 επίσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτές οι αρχές επίσης υπάρχουν ε, στην χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο Ένωσης, ε, οδηγία 2178 για την κατάρριξη της διακριτικής μεταχείρισης στην εργασία λόγω σεξουαλικών πεπιθήσεων ηλικία ε, ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Πέρσι υπέβαλε η Επιτροπή μία πρόταση για να διευρύνει αυτή την προστασία και σε άλλου τομεί. Ε, το Συμβούλιο συζητά, επεξεργάζεται αυτή την πρόταση και έχει εκδώσει ήδη θετικό δημοψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλωσορίζουμε αυτή την ε, πρωτοβουλία και ελπίζουμε ταχύτατα να εγκριθεί σε, αυτά συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο μπορούν φυσικά τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ε, νομοθεσίες υπό την προϋπόθεση, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το πρωτογενές και το δευτερογενές δίκαιο της Ένωσης. Και αυτό το κάνουν μόνο αν αποδείξουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούλιο εγκρίθηκε αυτή η νομοθεσία από τη Λιθουανική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, μία τροπολογία που τώρα συζητείται για την τροποποίηση του ποινικού δικαίου που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλε ανησυχίε στη Σουηδική Προεδρία. Ακόμη δεν έχει αρχίσει να ισχύει. Ο στόχο είναι η απαγόρευση ε, τη προώθηση ενό συγκεκριμένου σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό σημαίνει παραβίαση των θεμελιωδών αξιών, τη ελευθερία έκφραση και τη ισότητα όλων των ανθρώπων. Και εμεί επανειλημμένα έχουμε διευκρινίσει Πια ποια είναι η θέση μας σε επαφές με τη λιθουανική κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να Αναφέρουμε εδώ ότι δεν έχει επίσημο ρόλο σε αυτό το τομέα το Συμβούλιο. Γιατί ε, δεν είναι θέμα Συμβουλίου ε, το αν συμμορφώνεται μια εθνική νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο. Το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κρίνει αν πληρούνται οι εθνικές υποχρεώσεις δυνάμει της ε, συνθήκης. Ε, και αυτό δεν ε, καλύπτει μόνο την παρακολούθηση σωστή σωστής μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία και υλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά έχει σχέση και με την τήρηση του πρωτογενούς δικαίου των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκινήσει διαδικασίες για ε, παραβίαση των συνθήκων αν κρίνει ότι παραβιάζονται από κάποιο κράτος μέλος. Για το άρθρο 13 της συνθήκης ε, για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα το Συμβούλιο θα δήλωνε αποτροπιασμό αν ε, διαπίστωνε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, εθνοτικής προέλευσης, ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων, αναπηριών, αλλά χρειάζεται και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Βάσει του άρθρου 7 της ε, συνθήκης, ε, θα πρέπει ή η πρόταση, να υπάρξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μία πρόταση από το 1 τρίτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Σας ε, καθησυχάζω. Ε, αποτελεί προτεραιότητα για μας ε, το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης των ομοφιλοφιλών ε, και εξάλλου διοργανώνουμε και μία σχετική σύσκεψη στην Στοκόλμη... στις 16 με 17 Νοεμβρίου. Πιστέψτε με, παίρνουμε στα σοβαρά τις ανησυχίες για γιατί πρόκειται για τη ρίση των θεμελιωδών ελευθεριών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να κινηθούμε στο εφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ε, ε κοινοποίησα τη θέση μας, σας ανακοίνωσα και ποιοι είναι οι περιορισμοί. Δεν μπορούμε να κινηθούμε από μόνοι μας. Σας ευχαριστούμε πάντως για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το ζήτημα. Al Ευχαριστώ Υπουργέ, ο λόγος στον ε, Επίτροπο Μπαρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Υπουργό ανέφερε πολύ σωστά και πλήρως ε, τη νομική πτυχή αυτού του θέματος. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κομισιόν Πολάκης έχει αναφέρει ότι καταδικάζει ρητά κάθε έκφραση και έκφανση ομοφοβίας που αποτελεί κατάφορη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα επανέλαβε τη θέση αυτή στις 23 Απριλίου του 2007 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια όπου εγκρίθηκε το ψηφίσμα για την ομοφοβία στην Ευρώπη. για τους ε, τομείς ε, κοινοτικής αρμοδιότητας η Ένωση και τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο καλούνται να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι ε, μια απαρέγκλητη άρχη του κοινοτικού δικαίου. Το νομοσχέδιο αυτό προστασία των ανελίκων κατά τέτοιων ε, έργων ή δραστηριοτήτων είναι αντίθετο με το περιεχόμενο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για ε, το οπτικό ακουστικό υλικό. Ενημερώσαμε λοιπόν τις λιθωνικές αρχές ε, ακόμα και πριν την υιοθέτηση του νομοσχεδίου ότι ορισμένες διατάξεις αυτού του νόμου θα δημιουργούσαν πολύ σοβαρές ανησυχίες σε ό,τι αφορά το αν είναι σύμμορφα με το κοινοτικό δίκαιο και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, η έγκριση αυτού του νόμου στις 14 Ιουλίου δεν διασκέδασε τις ανησυχίες που είχαν και ε, είχαμε και εμείς, που είχε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, αλλά και εμείς διότι δεν γίνεται σεβαστή η αρχή της μη διάκρισης αλλά και των δικαιωμάτων των παιδιών ένα από τα οποία είναι η πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για την πνευματική τους ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, η Κομισιόν δεν θα διστάσει να λάβει ή οδήποτε κατάλληλο μέτρο για να διασφαλίσει τον σεβασμό του κοινοτικού δικαίου και βεβαίως των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Λιθουανία συστάθηκε μια ομάδα εργασίας πρωτοβουλία της κυρία Γκριμποσκάιτε, πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να γίνουν ε, τροπολογίες, τροποποιήσεις ε, επί του νόμου αυτού. Τροποποιήσεις, ε, τροπολογίες που θα υποβληθούν στα τέλη Οκτωβρίου στην Λιθουανική Βουλή. Η Κομισιόν οφείλει προφανώς να αναμείνει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτής της Επιτροπής και το περιεχόμενο των τροπολογιών που θα προτείνει για να μπορέσει να αποφανθεί οριστικά επί του νόμου ως θα τεθεί σε ισχύ στη Λιθουανία. Ως εκ τούτου, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μάλστρομ που είπε ότι η Κομισιόν είναι αυτή η οποία εποπτεύει την κατάσταση και ενδεχομένως θα προτείνει να επιβληθούν κυρώσεις κατά της χώρας λόγω μη συμμορφώσεις με το κοινοτικό δίκαιο και ως εκ τούτου των, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά ε, είχα να πω και νομίζω ότι η θέση μας είναι απόλυτα σαφής. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Στο όνομα των ομάδων τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι Λαντεσβέργης για δύο λεπτά. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε παρόλο που δεν έχει ισχύσει ακόμη προβλέπεται μόνο μία γραμμή όπου απαγορεύει ε, την ε, ομοφιλοφιλία για τους ανηλίκους. Είναι μία μονομένη ε, περίπτωση άρα θα πρέπει να υπάρξουν οι σχετικές τροπολογίες ενώ η δικιά μας, ε, το δικό μας ψήφισμα δημιουργεί ένα ολόκληρο θέμα διότι ε, για την ομοφιλοφιλία μεταξύ ανηλίκων ε, αναφερόμαστε μόνο σε ε, προώθηση για τους ανηλίκους και όχι σε ομοφιλοφιλία. Η προώθηση είναι κάτι παραπάνω από την ε, απλή ε, εκπαίδευση και θα πρέπει να περιέχει και κάποια ανοχή στο κάλεσμα των ομοφιλοφίλων ενώ προώθηση προς την ομοφιλοφιλία μπορεί να σημαίνει κάτι παραπάνω δηλαδή ε, να ε, ε, επιστρατευτούν οι ανήλικοι και να ξεκινήσουν πορνεία των ανηλίκων. Ε, γι' αυτό θα παρακαλούσα τώρα να εξετάσετε συνάδελφοι αν εσείς θα θέλατε να δεχθείτε όλες αυτές τις προκλήσεις για τα παιδιά σας. Ίσως κάποιος μπορεί αλλά τι θα γίνει όμως ε, υπάρξει ε, συνεχής τέτοια παρενόχληση οπότε ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και το δικαίωμα των παιδιών ε, να μην βιάζονται πνευματικά και να προστατεύονται από οποιαδήποτε παρεκτροπή. Προτείνω λοιπόν να ε, στηρίξουμε τις θέσεις που θυμίζουν σε όλους τα δικαιώματα των παιδιών και να διαγράψουμε την παράγραφο 1 που δεν έχει καμία δουλειά σε αυτό το σημείο. Ε, παρακαλώ να ε, ακολουθήσουμε τα υψηλά ιδεώδη της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Μωράες mr landsbergis Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Λανσμπέργκη δεν μα έπεισε με την αιτιολόγηση αυτή τη νομοθεσία. Με ξάφνιασε. Νόμιζα θα τα κατάφερνε καλύτερα. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασαν τη βαθύτατη ανησυχία. Αυτή είναι η σωστή γραμμή. Η κατάργηση τη διακριτική μεταχείριση και η ελευθερία έκφραση είναι θεμελιώδει απαραίτητε αρχέ των ευρωπαϊκών νόμων στη χώρα μου. Το 88 είχαμε μια τέτοια ε, νομοθεσία, αλλά τώρα είναι ιστορία κατά καταργήθηκε και το ίδιο θα συμβεί και ε, με αυτόν γιατί οι κοινέ αξίε μα είναι και η δύναμή μα. Η κοινή προσπάθεια να προστατεύουμε τι θεμελιώδει ελευθερίε ε, των πολιτών μα. είναι πάντοτε δύσκολο όταν ε, όλοι κατηγορούν μία χώρα για μία, επειδή όλοι ισχυρίζονται ότι παραβιάζει αυτέ τις κοινέ αρχέ. Αλλά μπορούμε να αναλύσουμε ποιε είναι αυτέ οι κοινέ αρχές γιατί η κατάσταση όπω είπε η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι ανησυχητική. Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να επιτελέσει το καθήκον του και υπάρχει ε, πρόβλημα με τη, τέτοιου είδου νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ε, η το Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Λιθουανία να ε, καταδικάσει αυτόν τον νόμο και να περάσει στην ιστορία ε, στις ζωμαϊκές καλένδες. Ο κύριος Ντόνσκης ε, για δύο λεπτά. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η νομοθεσία στη Λιθουανία σχετικά με την προστασία των ανηλίκων είναι πολύ αντιδημοκρατικός. Τονίζω ότι ο νόμος αυτός έχει υποβληθεί δύο φορές από τον πρόεδρο της Λιθουανίας αλλά περίφθη από το Κοινοβούλιο και τα μέτρα αυτά είχαν ε, ε, επίσης κατακριθεί από τον τωρινό πρόεδρο Κρυμποσκάιτε πέραν ε, των ε, οργανώσεων προασπίσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι έχει ε, πολλές πολιτικές επιπτώσεις όπως η λογοκρισία και η αυτολογοκλησία διότι αντί να προστατεύσει τα παιδιά στρέφεται κατά των ομοφιλοφίλων πολιτών της χώρας και ε, ε, η αναγνώριση ορισμένων εκτρόπων ε, είναι σαφώς απορριπταία αλλά στην αρχές του 21ου αιώνα δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια νομοθεσία την οποία θεωρούμε σαν μια τυχή κίνηση και σαφή παρανόηση διότι λαμβάνοντας υπόψη ε, ότι ε, ε, συζητούνται ποινικέ ρήτρε της νομοθεσίας για την απαγόρευση της ομοφιλοφιλίας και των εκφράσεών της σε δημόσιους χώρους και αν αυτό δεν είναι καταπίεση των πολιτών τότε τι είναι. Ο νόμος αυτός είναι απαράδεκτος αλλά προσπαθεί ουσιαστικά να να καταπιέσει το λαό και γι' αυτό στηρίζω το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέντα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική αυτή η καμπή στην ιστορία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτή τη συζήτηση δεν θα την ε, κάναμε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Κανένα κοινοβούλιο δεν θα διανοεί το να περάσει ένα τέτοιο νόμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ε, θέμα που αφορά τη Λιθουανία, τα εσωτερικά της Λιθουανίας. Είναι ένα θέμα που αφορά την ευρωπαϊκή αξιοπιστία στο σύνολό της. Το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να σιωπήσει ενώ σε χώρα μέλος εγκρίνονται νόμοι που καταπατούν τέτοια και τόσα θεμελιώδη ε, δικαιώματα και διακριτικές ε, και επιβάλλονται διακριτικές ε, μεταχειρήσεις. Η αμφιφιλία, η αμφιλοφιλία, η ομοφιλοφιλία είναι θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο κύριε Λαντσμπέργκης δεν είναι ταμπού. Πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για αυτά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζητούμε την καταπάτηση των στερεοτύπων. Είναι μια κανονική συζήτηση που γίνεται χωρίς απαγορεύσεις και χωρίς ε, σκιάχτρα. Ευχαριστώ. Σημάσκι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο λιθονικός αυτός νόμος για την προστασία των ανηλίκων πηγάζει από ανησυχίες που υπάρχουν ε, και την επιθυμία να προστατεύσουν τευθούν οι ανήλικοι από διάφορους ε, κινδύνους. Το ζητάνε οι γονείς αυτών των παιδιών. Όλοι θα συμφωνήσετε ότι πρόκειται για ένα επίγον πρόβλημα. Και αυτές είναι οι προθέσεις μας και άρα θα, ε, πρέπει, θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές ε, και όχι να επικρίνονται. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτό δεν έχει καμία επιρροή επί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όλα τα ζητήματα που τίθενται μέσα στην προφορική αυτή ερώτηση σχετίζονται με την εθνική νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει καμία αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Δεν καταλαβαίνω καν γιατί συζητείτε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ε, υπάρχει αυτή η υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα σχέδια ψηφίσματος που έχουν ε, υποβληθεί. Ε, ένα λεπτό, Σπένσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα δεν μιλάμε εδώ για ιδεολογία. Μιλάμε για την ισότητα των ανθρώπων. Ευχαριστώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, έλαβαν σαφώς θέση αυτή τη φορά η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ελπίζουν να κινηθούν τώρα από κοινού όταν διαπιστώνουμε παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών. Μιλάμε για την τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Ότι οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι παράνομη. Φανταστείτε να απογορευτεί το να αγωνιζόμαστε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου και του γενετησίου προσανατολισμού. Δεν χρειάζεται να απαριθμίσω τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζει αυτό το νομοσχέδιο. Απλά θέλω να δηλώσω τη ρητή υποστήριξή μου για το ψήφισμα. Ελπίζω ομόθυμα, σύσσωμο το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οι υπόλοιποι ομιλητέ ε, θα πάρουν το λόγο τώρα. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης. Σε δύο λεπτά ο κύριος Ματιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, και κυρία Μάτια. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και όλους τους συναδέλφους η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεως και ιδίω όσε αναφέρονται στις σεξουαλικές, στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο στη Λιθουανία που δημιουργεί τόσα προβλήματα ώστε ασχολήθηκε η κυρία Κρυποσκάιτε έθεσε βέτο και ε, ε, σε μια ομάδα εργατίες η οποία θα υποβάλει τροπολογίες. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι το πρόβλημα θα λυθεί και το κράτος μέλος θα μπορέσει να λύσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί μια διάκριση κατά των σεξουαλικών προσανατολισμών. Ορισμένοι πρότειναν ένα ψήφισμα και ευτυχώς μπορέσαμε να βρούμε μία, ένα κοινό ψήφισμα. Ελπίζω λοιπόν συνάδελφοι ότι αύριο το ψήφισμα θα υπερψηφιστεί, το πρόβλημα θα λυθεί. Είναι προφανές, ε, προφανώς σημαντικό η πνευματική και... Ε, ε, ε, η υγεία των παιδιών να προστατεύεται αλλά έχουμε ένα γραφείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα το ε, παλέψαμε για να καταρτιστεί άρα τώρα δεν θα την αγνοήσουμε παρακαλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε το κοινό ψήφισμα ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και ελπίζω ότι ότι και στο, στην Ολομέλεια αύριο θα υπερψηφιστεί. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ε, ε, η κυρία Λιντσοβικούτε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, πρωτοβουλία να αναλάβει το θέμα ε, ε, αυτό διότι στην χώρα μου είναι μια παραβίαση του δικαιώματος για πληροφόρηση και κακώς το θέμα αυτό προτάθηκε στη Λιθουανία χωρίς να έχει επαληθευτεί. Υπάρχουν διάφορες α, ε, α, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες προειδοποίησαν αλλά εις ε, Θα, ε, ε, αυτό οδήγησε σε διαφορές μεταξύ των ομάδων της κοινωνίας και η λιγενινή πρόεδρος έχει θέσει βέτο κατά αυτού του νόμου, κατήρτισε μία ομάδα εργασίας και θα συζητηθούν τα πορίσματα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ελπίζουμε ότι η νομοθεσία θα βελτιωθεί και ε, ε, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία σύγχρονη νομοθεσία. Πριν έξι χρόνια οι σοσιαλδημοκράτες είχαν ε, ψηφίσει ε, μία, ε, ένα νόμο για την ίση μεταχείριση σε όλους τους τομείς της ζωής και συζητήσει και από το Συμβούλιο. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα θα έπρεπε να ενθαρρύνει την χώρα αυτή να υπερψηφίσει τα θεμελιωδή δικαιώματα του ανθρώπου αλλά σύμφωνα με ε, το σύνταγμα της χώρας. Η κυρία Μπούτσο για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, ε, μου με σοκάρει το ότι ένα τέτοιο κοινοβούλιο όχι μόνο προτείνει αλλά και ψηφίζει τέτοια μέτρα το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και στη Λιθουανία και σε όλη την Ευρώπη λες και ήταν κάτι ε, για το οποίο θα πρέπει να ντρέπονται και θα πρέπει κανείς να προστατεύσει τα παιδιά ε, ενώ πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση στην Ευρώπη είναι θέματα τα οποία έτυχαν διαπραγματεύσεων και ε, γι' αυτό τώρα θα ήθελα να επανέλθω στη διαβεβαίωση του Επιτρόπου που είπε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προτού ψηφιστεί. Κυρία Νικολάζη, στη διαδικασία κάτσε για ένα λεπτό. Ο κύριος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υιοθέτησε η Λιθουανία ένα νόμο με στόχο την προστασία των παιδιών και των ανηλίκων κατά πληροφοριών που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά ε, το μέλλον τους. Η κοινωνική πολιτική, ισχυρίζονται κάποιοι, είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και άρα δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρχουν επικρίσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάμε για διεθνή πρότυπα. Εγώ ε, εξέτασα όλη αυτή την επιχειρηματολογία και συμφωνώ, θεωρώ, ότι αντίθετα ενισχύει την προστασία των παιδιών. Δεν χρειάζεται να εκτίθεται σε πληροφόρηση και σε ε, εικόνες που ε, από τις οποίες ε, θέλουν να τους ε, προστατεύσουν οι γονείς τους. Παραβιάζεται εδώ η αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο της συνθήκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για τις οικογένειες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ε, grazie, ένα λεπτό. Ε, πρόεδρε, πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούνται δράσεις ε, και ενέργειες της λιθουανικής κυβέρνησης με αρνητικό τρόπο. Οι συντάκτες ε, του νομοσχεδίου είχαν κάποιες συγκεκριμένε επιθυμίες και προθέσεις αλλά το νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν στον 21ο αιώνα. Η λιθουανική κυβέρνηση είναι πεπισμένη για την αντικειμενικότητα και την αξία του νομοσχεδίου. Βλέπουμε την ισχυρή ενθερμό αντίδραση της Επιτροπής και του Συμβουλίου κατά της ενέργειας της λιθουανικής ε, κυβέρνηση Μας λένε δεν πρέπει να καρκινοβατούμε και να περάσουμε ξανά στο μεσαίο. Να Πρέπει να σεβόμαστε την ευρωπαϊκή παράδοση. Χρειάζεται και η συζήτηση, χρειάζεται και το ψήφισμα για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Βίκστρομ, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Όλοι γεννιόμαστε ίσοι και υπάρχουν αρχές που δεν πρέπει να παραβιάζονται. Πρέπει σαφώς να περάσουμε το μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα ε, των ανθρώπων ανεξάρτητα από τη χώρα την οποία συζητάμε. Η ελευθερία έκφρασης, ε, ανοχή, άνεξη, αυτές είναι οι αξίες μας. Ε, ξεκαθάρισε η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι θα υπάρχει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που θα καλύπτει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόεδρε, διαπιστώνουμε με λύπη σήμερα ότι η Λιθουανία που έχει ζήσει τη δικτατορία, ε, την ε, καταπίεση και που έγινε μια ελεύθερη χώρα, τώρα παραβιάζει την ελευθερία και δείχνει παντελή έλλειψη ανοχής. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές ε, αξίες. Με πυγμή πρέπει να στιγματίσουμε τον νόμο. Αύριο πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η βασικότερη ευρωπαϊκή αρχή είναι η αγάπη. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμπόσκα για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ και η Σλοβακία είχε καταδικαστεί γιατί, ε, για μια παρεμφερή νομοθεσία η οποία προσπαθούσε να ε, ε, να προστατεύσει τα παιδιά από την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση της κοινωνίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, ζητάτε εδώ να ε, υπερισχύσει ε, και να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Οργάνωση που δεν έχει δικαίωμα να ε, επέμβει σε, σε μια εθνική νομοθεσία. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κατακριθούν και εδώ ορισμένες νομοθεσίες οι οποίες ε, ε, δεν σέβονται το δικαίωμα της ποικιλομορφίας και το δικαίωμα οι γονείς να αναθρέφουν τα παιδιά τους όπως θέλουν. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην Υπουργό κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι σαφές πως τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, συμφωνούν ε, σε αυτή τη συζήτηση. Ε, δηλαδή, ανοχή να καταδικάσουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης και της κατάργησης διακριτικής μεταχείρισης λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού. Τα κράτη-μέλη φέρουν την ευθύνη να σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες και τη κοινοτική νομοθεσία που ισχύει σε αυτό το τομέα. Και νιώθουμε βαθύτατη ανησυχία για αυτό το ζήτημα και ξέρουμε ότι υπάρχουν επικρίσεις και στην ίδια τη Λιθουανία. Η πρόεδρος ε, Γκριμπάους Κάιτε που ε, διατέλεσε και επίτροπος έχει μιλήσει για την ανάγκη προστασία ε, ε, προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και έχει κινήσει από μόνη της την διαδικασία για να διερευνηθεί το ζήτημα και να ληφθούν οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες. Και θα Ελπίζουμε ότι με αυτέ τι κινήσει και τι δικέ μα πρωτοβουλίε τελικά δεν θα τεθεί σε ισχύ αυτό το νομοσχέδιο. Σα ευχαριστούμε, ο Επίτροπο Μπαρό. Συμφωνώ με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η κυρία Υπουργό και ελπίζω ότι η Επιτροπή που σύστησε η κυρία Αγκριβοσκάιτε θα δώσει την ε, δυνατότητα στην ε, Λιθωνική Βουλή να καταστήσει τον νόμο αυτό συμβατό και με το κοινοτικό δίκαιο. Και το λέω αυτό διότι ορισμένε διατάξει του νόμου φοβούμεθα ότι είναι αντίθετε ε, με το περιεχόμενο ορισμένων οδηγιών για τα απτικοακουστικά μέσα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για το οικογενειακό δίκαιο δεν έχουμε αποφανθεί ε, αρμοδιότηση των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, ό,τι ελέγχθη κατά τη διάρκεια της συζήτησης καταδεικνύει ότι θα πρέπει να μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος ε, τα πράγματα και ιδιαίτερα η Λιθουανία να το κάνει αυτό και θα το κάνει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έλαβα πέντε προτάσεις ψηφίσματος. Η συζήτηση ε, Ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο.